facciamo finire la telefonata al nostro Καλημέρα σας συνάδελφοι. Παρόλο που είμαστε σε περιορισμένη σύνθεση, επειδή είναι παρόντες όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν τις ψηφοφορίες θα προεδρεύσω εγώ και μετά θα αναλάβει ο κύριος Μπούζεκ για να συνεχίσουμε την διεκπαιρέωση μερίσεις διάταξη που είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Ανακοινώσει του Προέδρου, καταρχήν έγκριση μερίσης διάταξης και ε, βλέπω να μην υπάρχουν προβλήματα και μετά τις θερινές διακοπές έχουμε το πρόγραμμα των συνεδριάσεων. Έχουμε πολύ φορτωμένο νομοθετικό πρόγραμμα, ειδικά στη δική μας Επιτροπή. Γι' αυτό κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιήσουμε κάπως το χρονοδιάγραμμά μας. Γι' αυτό και σας προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Φυσικά θα ακολουθήσει και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και γραπτά υπομνήματα με τις αλλαγές. Οπότε μετά τις θερινές διακοπές 4 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες το απόγευμα, αυτή είναι μια ήδη προγραμματισμένη συνεδρίαση, 11 Σεπτεμβρίου έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 7 με 8.30 το βράδυ και μετά για την ε, διακυβέρνηση, για την ενέργεια και για την Επιτροπή. Και έπειτα μόνο η Επιτροπή Ήτρε από τις 20 και 30 μέχρι τις 22 και 30. Και στις 2 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο θα έχουμε συνεδρίαση από τις 19 μέχρι τις 22 και 30. Όπως βλέπετε το φθινόπωρο θα είναι αρκετά και όπως σας είπα, όλα αυτά τα σημεία θα σας τα στείλουμε και γραπτός. Νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεών μας και περνάμε στην εξέταση της το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης πρόκειται για τον ε, σεβασμό, μάλλον για τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή ε, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το σεβασμό της ε, ιδιωτικής ζωής καθώς και την προστασία των προσωπικών στοιχείων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο κατάργας στην κυρία Κάλλας που είναι η συγγέντριά μας Νομίζω ότι θα μιλήσει για 5 με 6 λεπτά και έπειτα θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους συνάδελφους. Παρακαλώ κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Όπως επισημάνατε, κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε το θέμα του χρονοδιαγράμματος, το επισήμανα και σκιώδης ηγητές, γι' αυτό και προτείναμε ε, και παράταση της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών και αναβολή. Ε, δεν συμφωνώ με αυτή την ε, παράταση, γιατί πριν από ένα μήνα έχει στέλνει το θέμα για μετάφραση. Οπότε δεν συμφωνώ με την παράταση του χρονοδιαγράμματο ε, για τη διεκπαιρέωση τη έκθεση. Και επειδή και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών παρέμεινε στο πρόγραμμά τη, θα πρέπει και εμεί να τηρήσουμε το δικό μα χρονοδιάγραμμα, αν θέλουμε να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αυτά ω προ τη διαδικασία, ω προ την ουσία και το πεδίο εφαρμογή. Δεν τροποποιήθηκαν οι ορισμοί, έμειναν στου ορισμού του κώδικα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών πρότεινε τη συμπερίληψη ορισμών στην οδηγία για την ιδιωτική ζωή στην ηλεκτρονική σφαίρα, η privacy. Επίσης, ε, θέλω να προστατεύσω την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών, αφήνοντας όμως ελεύθερο το περιθώριο για την καινοτομία. Πολύ συχνά ε, συζήτηση περιγράφεται μονοσήμαντα, σαν είναι άσπρο-μαύρο. Αν όμως χάσουν οι πάροχοι ε, της, την εμπιστοσύνη, οι τελικοί χρήστες για την κατάχρηση των δεδομένων τους, ε, θα χαθεί η εμπιστοσύνη. Και μερικές φορές προτείνουμε περισσότερη καινοτομία, ε, συμπεριλαμβάνοντας το, το στοιχείο του συμβατού σκοπού για την επεξεργασία των δεδομένων με βάση το GDPR και ε, την περίπτωση της εξαίρεσης ε, όπου απαιτείται η, η συγκατάθεση του τελικού χρήστη της υπηρεσίας. Πάντως, σε η γνωμοδότησή μου τάσεται υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο για την Επιτροπή είναι να γίνει ουδέτερη από τεχνολογική άποψη η πρότασή μας. Για παράδειγμα, επικεντρωνόμαστε, η Επιτροπή επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους φιλομετρητές, στους browsers ενώ όλο και ε, περισσότερη έμφαση δίνεται στις συσκευέ που χρησιμοποιούν εφαρμογές και άλλες. Επίσης γίνεται διάκριση μεταξύ των cookies ε, του ίδιου και του τρίτου μέρους. έχουν κάποια, κάποια επιρροή στην ιδιωτικότητα. Μερικά cookies χρειάζονται για την βελτίωση της υπηρεσίας ή για την παράδοση της υπηρεσίας, την παροχή της υπηρεσίας. Και ενώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις εταιρείε για να συνεργάζονται και να προτείνουν πρακτικές και εύχριστες λύσεις, θέλω να υπάρχει και δυνατότητα επιλογής για το χρήστη. Αν ο χρήστης ε, δεν δώσει τη συγκατάθεσή του και μετά δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες, αυτό δεν είναι, να έχει, δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρεωμένο δηλαδή είτε να δεχτεί τα κούκκι και να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, είτε να τα απορρίψει και να μην έχει πρόσβαση. Αυτό δεν είναι επιλογή. Η πραγματική επιλογή έγκυται στο ότι μπορεί να παρακολουθεί τα πράγματα. Επίσης, ε, ε, τι είδους ε, δεδομένα μπορεί ο χρήστης να μοιράζεται και με ποιον, να ανταλλάσσει. Θέλουμε καλύτερη σχέση εμπιστοσύνη εταιριών, παρόχων, υπηρεσιών και χρηστών και να μπορούν οι χρήστες να χαρακτηρίζουν, να δουν ποια είναι τα πιο ευαίσθητα στοιχεία. Και επίσης να δώσουμε πιο φιλικές προς το χρήστη λύσεις ε, για το tracking, για την παρακολούθηση των στοιχείων. Γιατί να μην, γιατί να μπορούν να ρωτούν οι εταιρείε στον χρήστη τι είδου ε, πληροφορίε χρειάζεται. Επίση, η συγκέντρωση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε λάθο ε, ω προ τη διαφήμιση και να κάμψει την εμπιστοσύνη του χρήστη προς τον πάροχο. Επίσης, στο θέμα της επιλογής, έχω κάποιες αμφιβολίες ό,τι αφορά την περίπτωση του, της παρακολούθησης με ασύρματο δίκτυο. Αυτό δεν δίνει επιλογές και ίσως είναι αντιπαραγωγικό και δημιουργήσει άγχος στους πολίτες, γιατί όταν βλέπουν ότι παρακολουθούνται δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, απλώς βλέπουν την κοινοποίηση. Οπότε καλύτερα να περιορίσουμε το Wi-Fi tracking μόνο για στατιστικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τα public directories, ε, μερικές φορές τα στοιχεία δεν ε, συγκεντρώνονται από δημόσιους φορείς, από εταιρείε τηλεπικοινωνιών, οπότε είναι ίσως δύσκολο να πετύχουν τη συγκατάθεση. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, πρότεινα διαγραφή του άρθρου γιατί θεωρώ ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ του άρθρου 40 τις οδηγίε για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το GDPR, τους γενικού κανονισμούς και τη συγκεκριμένη οδηγία, ήδη αυτά τα θέματα καλύπτονται. Τέλο θεωρώ ότι το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 11, που δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη ε, να έχουν πρόσβαση σε επικοινωνίε ε, σε μηνύματα των πολιτών, είναι υπερβολικά γενικό το πεδίο εφαρμογή. Ε, η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οδηγία e-privacy είναι υπέρ της ιδιωτικότητας ε, και του ελέγχου του πολίτη για τα θέματα της ειδικής του σφαίρας. Οπότε παραπέμπω στην οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Επίσης, τα κράτη-μέρη μπορούν να μην επιβάλλουν ε, υποχρεώσεις που μειώνει την ασφάλεια των ε, υπηρεσιών επικοινωνιών. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαραγωγικό. Γιατί από τη μια έχουμε πολλούς κανόνες για, την, για τις εταιρείε για να προσπίσουμε την εμπιστευτικότητα και μετά προβλέπουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη όποτε θέλουν να ζητούν από τις εταιρείε να υποβαθμίσουν αυτές τις προδιαγραφές. Αυτά ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ κυρία Κάλλας γιατί ήσασταν σαφέστατοι και σεβαστήκατε και το χρόνο ομιλία σας. Πρώτη παρέμβαση, αντικατάσταση του συναδέλφου Μπόνι από τον συνάδελφο Ρούμπι. Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο Κάγια Κάλλας γιατί νομίζω ότι πολύ σωστά παρουσιάζει τα θέματα για το πώς αυτόν τον εικονικό κλάδο θα έχουμε μία αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου. Οι νέοι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξουν μεγάλο ρόλο και θα συλλέγονται πολύ μαζικά στοιχεία. Οπότε το θέμα της ιδιοκτησίας τους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση όχι μόνο της ιδιωτικής σφαίρας αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά ακριβώ ε, την ε, ιδιωτική σφαίρα, να φροντίσουμε ούτω ώστε ε, κάποια στοιχεία να μην είναι κρυπτογραφημένα για να μπορούν να συλλέγονται για στατιστικούς στόχους, αλλά μόνο για τέτοιους λόγους. Μόνο εφόσον έχει έννοια. Και φυσικά είναι επίσης σαφές ότι πρέπει να εγγυηθούμε την τεχνολογική ουδετερότητα και την διαλειτουργικότητα Αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους καταναλωτές. Και επίσης η διαφάνεια. Για παράδειγμα, πώς λειτουργούν τα κούκι. Γιατί μπορούν ε, να προκύψουν και από ιδιώτες. Πρέπει να γνωρίζουν ποια στοιχεία περιλαμβάνονται. Έχουμε στην Αμερική νέες πανεπιστημιακές σπουδές που ασχολούνται με το ποια στοιχεία αξιοποιούνται καθημερινά από τους προσωπικούς μας υπολογιστές. Οπότε <clears throat> είναι αποφασιστικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην προκύψει επιπλέον ε, γραφειοκρατία. Ξέρουμε ότι ο υπεφορτισμένος με την ασφάλεια των δεδομένων και όλες ε, οι εντολές του σημαίνουν συμπληρωματική γραφειοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να ξέρουν τι πρέπει να αναλάβουν. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα την εισηγήτρια, διότι η έκθεσή της ε, προσπαθεί όντως ε, να είναι ισορροπημένη. Ξέρουμε ποιος είναι ο βασικός κανονισμός και η οδηγία η οποία συζητιέται τους τελευταίους μήνες. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής κρυπτογράφηση όταν αποστέλει ένα μήνυμα από το α στο β. Πρέπει λοιπόν να σώσουμε τις παλιές αξίες μέσα στις νέες τεχνολογίες. Και πρέπει λοιπόν να εξαγάγουμε και τα διδάγματα από την χρήση αυτών των τεχνολογιών στο παρελθόν. Δηλαδή και οι νέες αυτές τεχνολογίες πρέπει να εξασφαλίσουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ σωστής χρήσης και της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας, να ξέρουμε πώς ταξιδεύουν τα, τα δεδομένα, συγγνώμη, ποιες αυτόματες ε, ανταλλαγές ε, στοιχείων Πρέπει να φτιάξουμε μια νέα εταιρική σχέση του κοινού με τους ιδιωτικούς φορείς, ούτω ώστε όλα αυτά τα νέα δεδομένα να είναι σαφές πώς αξιοποιούνται, γιατί όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Κουρουμπάσεχ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη θαυμάσια εργασία της για το θέμα αυτό. Πολύ σωστή βάση και αντικειμενική βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι καλό που είναι και από την Εστονία που είναι πραγματικά πρωτοπόρα στην ψηφιακή τεχνολογία. Βεβαίως ένα βασικό θέμα είναι η παρακολούθηση και τα κούκκι. Πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των κούκκι που είναι απόλυτα αναγκαία για τη λειτουργία του δικτύου και του site και των άλλων. Έχουμε τα κούκκι απόδοσης και τα λειτουργικά κούκκι. Αυτά είναι τα μεν και από την άλλη μετά είναι τα διαφημιστικά ή τα κούκι που στοχεύουν ε, τους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς κανόνες που να δίνουν επιλογές από την αρχή, μέσω του σχεδιασμού, μέσω των ρυθμίσεων, μέσω των οποίων ε, ο καταναλωτής ε, μπαίνει στο ίντερνετ. Πρέπει να σταματήσουμε κάποιες πρακτικές. Δεν μπορούν να αποδεχθούν Συγγνώμη, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πρακτική που απαγορεύει στου χρήστε να μπουν σε ένα site μέχρι να αποδεχτούν τα κούκκι. Αυτό είναι ιδιαίτερα βλαβερό. Ένα άλλο τομέα που είναι πολύ σημαντικό είναι η περιοχή όπου δεν θα υπάρχει συνένεση. Για παράδειγμα, για κάποια πράγματα, για κάποια δίκτυα, για να βλέπουμε τις ροές θερμότητας. Βεβαίως η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι με ανώνυμη ή ψευδανώνυμη μορφή αλλά πρέπει να μπορεί να συλλεγεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό εννοώ τομέας όπου δεν πρέπει να υπάρχει συνένεση. Ένα άλλο θέμα. Η παρακολούθηση του Wi-Fi, όπως λέει η πρόταση Επιτροπής, θα πρέπει να αναφέρεται ε, ε, σε ένα σήμα η περιοχή όπου υπάρχει αυτό το Wi-Fi tracking και πρέπει θα να φαίνεται αυτό και σε αυτά τα οποία βλέπει ο καταναλωτής όταν χειρίζεται τους υπολογιστέ του. Αλλά θα πρέπει για παράδειγμα να υπάρχει δυνατότητα να, τηλεφωνη... να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες επίγουσας ανάγκης οι χρήστες. Το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την επεξεργασία των μεταδεδομένων. Πρέπει να επιτρέπεται σε κάποιες περιπτώσεις. Για την ασφάλεια. Ζωτικό είναι μέσω του κανονισμού να δούμε πώς θα γίνεται η επιστοποίηση των, ε, του εξοπλισμού τερματικών. Όχι να είναι υποχρεωτικό, να ξεκινήσει η διαδικασία. Υπάρχει σαφής ανάγκη για προδιαγραφές ασφαλείας για τα τερματικά, όπως για παράδειγμα η σήμανση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση για το επίπεδο ασφάλειας ε, της κάθε συσκευή. Επειδή υπάρχουν ε, πολύ περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις και προσπάθειες hacking, θα προτείνω κάποιες αλλαγές στο κείμενο για να ενθαρρύσουμε τις εταιρείες καταναλωτών να αναπτύξουν μηχανισμούς ασφαλείας για να, να ελέγχουν το περιεχόμενο. Όταν περνάνε τις γραμμές τους, για να αποφεύγονται αυτές οι επιθέσεις hacking ή, ή, e e e, τα, ή όταν φτάνουν στον τελικό καταναλωτή. Βεβαίω αυτό σημαίνει παραπάνω δουλειά για τι εταιρείε Telecom, αλλά είναι πολύ σημαντικό να σταματάμε αυτέ τι επιθέσει πριν φτάσουν στο χρήστη. Και συμφωνώ με τι ανησυχίε για το άρθρο 11, γιατί μπορώ να φανταστώ τι επινοήσεις μπορεί να προκύψουν στα 28 κοινοβούλια που θα εφαρμόσουν ενδεχομένω με διαφορετικό τρόπο αυτό το κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας τομέας που να μην μπορεί να φύγει. Και το τελευταίο τώρα είναι η, σειρά με την οποία θα γίνουν όλα αυτά. Δεν πειράζει αν γίνει αυτός ο κανονισμός 3-6 ε, μήνες μετά το GDPR. Αυτή πρέπει να είναι η εντολή του, της Επιτροπής, ε, οριζόντια, αλλά και του Κοινοβουλίου. Ναι. Είμαστε λίγοι έτσι κι αλλιώς, ε, λίγο ξεφύγαμε από το χρόνο μας, ε, αλλά δεν είμαστε πολλοί, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο large. Οι υπόλοιποι δεν τους βλέπω. Ναι, να δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Κέλλη που το ζήτησε. Θεωρητικός για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Μάλιστα, θεωρητικό. Καταρχάς να ευχαριστήσω την συγγήτρια, την κυρία Κάλλα, για την παρουσίαση αυτής της νομοδότηση. Ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να βελτιώσει την ποιότητα των επικοινωνιών, να ενημερώσει τους ε, κανόνες αλλά δεν θα πρέπει να μην ξεχνάμε και την ελεύθερη ροή των δεδομένων, που είναι άλλος στόχος. Πρώτα γενικά σχόλια. Στις 25 ε, μάλλον το, 2018 θα αρχίσει να ισχύει κανονικά αυτός ο κανονισμός και το GDPR και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν από τεχνολογικής άποψης να προσαρμοστούν στις ε, τεχνολογικές προδιαγραφές μετά από την έναρξη, μάλλον πριν την έναρξη ισχύω ε, του κανονισμού θα πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε αυτή την ημερομηνία. Η εισηγήτρια θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι σύμμορφη προς τον κώδικα τηλεπικοινωνιών και ο συζητητής για το GDPR πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση και συντονισμός με αυτό. Η πρόταση αυτή θέλει να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των, της επικοινωνίας, σε πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, η συγκήτρια ε, προτείνει ότι οι τεχνολογίες, ε, μάλλον ότι οι δικές της προτάσεις θα είναι ουδέτερες από τεχνολογικές άποψης. Ε, είναι πολύ καλύτερο, συμφωνώ, να εστιάσουμε στα pop-ups και όχι στα cookies, ώστε ο χρήστης να είναι ενήμερος για το τι συμβαίνει με τα δεδομένα του και να μπορεί να προβαίνει σε, σε επιλογές του όντας ενήμερος. Είναι Πιστεύω, νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε μια εξαίρεση για την ασφάλεια στην πρόταση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν γνωρίζουμε τη σημασία, τη διαστάσεις έχει πάρει το θέμα της ασφάλειας. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης για τα big data και για τις ε, φιλικές προς τους ε, χρήστες ε, λύσεις θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι ώστε να υπάρχει χώρος για καινοτομία. Τέλος, θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε το άρθρο 2 της πρότασης και να, που μιλάει για περιορισμούς, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν ξεπερνάμε την απόφαση του δικαστηρίου. Και η κυρία Κάλλας τέλος ανέφερε την εμπιστοσύνη. Είναι η λέξη κλειδί που διαρκώς αναφερόταν όταν μιλήσαμε για το GDPR και επίσης ανέφερε τη σημασία των επιλογών για τον τελικό χρήστη. Τέλος να πω, όπως και ο Πολ ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτό θα μπορέσει να καλύψει και το μέλλον, ώστε να καλυφθεί και η τεχνητή ευφυΐα, γιατί είναι ένας τομέας όπου υπάρχουν διαρκώς ταχύτατες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο... Α, υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μπαρσέρο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει με ενθουσιασμό την γνωμοδότηση της κυρίας Κάλλας. Εκτιμούμε ιδιαίτερως την ε, διεξοδική και πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή της εμπεριστατωμένη και χαίρομαι που τηρεί και το χρονοδιάγραμμα που ναι μεν είναι πολύ βραχυπρόθεσμο αλλά παρόλα αυτά είναι εφικτό. Ε, για μας είναι πολύ σημαντικό η έγκριση της γνωμοδότησης να λάβει χώρα το Μάιο του 2018. Και ο Μάιος του 2018 ε, δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία είναι σημαντικό γιατί το Μάιο του 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Γενικό Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων, το GDPR, οπότε καλό είναι να είναι συμβατά. Βέβαια το e-privacy, η οδηγία αυτή, είναι λέξη specialis σε σχέση με το Γενικό Κανονισμό. Ο Γενικό Κανονισμός περιλαμβάνει γενικές αρχές για όλους που συνδέουν τα δεδομένα, από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ε, νοσοκομείο, ενώ το e-privacy αφορά μόνο τις τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, αλλά είναι θα πρέπει να είναι συμβατές ε, αυτές οι δύο νομοθετικές πράξεις. Γι' αυτό και έχει νόημα ε, να ξεκινήσουν από κοινού το Μάιο του 2018 και ο Γενικός Κανονισμός και η Οδηγία e-Privacy. Και γι' αυτό πιέσαμε κάπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έγκριση έγινε τον ε, ε, Ιανουάριο του 2017, 14 μήνες θα περάσουν δηλαδή ουσιαστικά μέχρι το Μάιο του 2018. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πιεστικό το πρόγραμμα, αλλά και εμείς πιεστήκαμε για να υποβάλουμε την πρόταση τον Ιανουάριο και να καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ως προς το περιεχόμενο τώρα, Εκτιμούμε ιδιαίτερος ε, το έργο σας και βλέπουμε πολλά κοινά σημεία. χαίρομαι επίσης για την υποστήριξή σας κάποια συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν, οι ορισμοί. Η κυρία Κάλλας κράτησε τους ορισμούς, ε, κάτι που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κάτι που είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι η κάλυψη των ότι της ε, παραμένει είναι σημαντικό, γιατί αυτά τα νέα εργαλεία, το Skype, το WhatsApp, ε, χρησιμοποιούνται σχεδόν το ίδιο με τα παραδοσιακά μέσα. Οπότε η εμπιστευτικότητα των ε, επικοινωνιών να εξασφαλίζεται και με τα νέα εργαλεία επικοινωνίας, όχι μόνο με τα παραδοσιακά. Επίσης, ε, χαιρόμαστε γιατί συμφωνείτε με την ε, αρχή της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών με συσταλτική ερμηνεία. Με περιορισμένη έννοια. Όπως είπε η κυρία Κάλλας, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ παρόχων και τελικών χρηστών και θα πρέπει η διεύλη να είναι ασφαλής, να μην μπορεί κανείς να παρεμβαίνει στην επικοινωνία. Τώρα, δύο σημεία στα οποία κάπως παρεκκλίνουμε. Γιατί, ρωτήσατε, κρατήσαμε κάποια προοπτική πολιτικής. Καταρχήν για την περαιτέρω επεξεργασία. Επί του παρόντος, από τη στιγμή που η τηλεπικοινωνία έχει προσφέρει την υπηρεσία, ο πάροχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, στη συνέχεια τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα για άλλους σκοπούς για σκοπούς δηλαδή που δεν αφορούν την παροχή της επικοινωνίας. Αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ε, κράτησε αυτόν τον περιορισμό. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει γίνει η επικοινωνία θα πρέπει η πληροφορία να διαγραφεί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω. Κρατήσαμε αυτόν τον περιορισμό γιατί έχουμε την αίσθηση και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Να παραμείνουν απόρριτα αυτά τα δεδομένα και ο φόβος ε, της ε, ε, αλλεπάλληλης επεξεργασίας θα υποσκάψει την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν το επιτρέπουμε. Επίσης, από τη στιγμή που επιτρέπουμε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, ουσιαστικά εξουδετερώνουμε τον κανόνα που υπάρχει, τη δυνατότητα διαγραφής, γιατί θα πρέπει να λάβει η χώρα η διαγραφή από τη στιγμή που τα δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για το billing. Και αν επιτρέψουμε συνέχιση της χρήσης, ουσιαστικά εκενώνουμε περιεχομένου ή εξουδετερώνουμε το λόγο ύπαρξης του κανόνα της διαγραφής. Γι' αυτό και δεν επιτρέπουμε την ε, περαιτέρω επεξεργασία. Δεύτερο θέμα, τεχνική ουδετερότητα. Συμφωνούμε με την κυρία Κάλλας ότι η πρόταση ίσως ε, φαίνεται να παραίνει εστιασμένη στα κούκκι, που είναι ένα είδος τεχνολογίας και ένα είδος παρακολούθησης, γιατί υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι παρακολούθησης, αλλά αυτό ισχύει ως προς τις αιτιολογικές σκέψεις που περιλαμβάνουν κάποια παραδείγματα των άρθρων και οι αιτιολογικές σκέψεις αναφέρονται στα κούκκι. Αλλά αναφέρεται και σε, αναφέρονται και σε άλλες τεχνικές παρακολούθησης, ως, ε, όπως τα δεκτυλικά αποτυπώματα στη συσκευή. Αλλά το θέμα είναι, μας ενδιαφέρει τεχνική ουδετερότητα και ίσως ε, στις αιτιολογικές σκέψεις αιτιολογικών επικεντρωνόμαστε στην ε, κρατούσα σήμερα τεχνολογία, αλλά μας ενδιαφέρει η τεχνική ουδετερότητα. Δηλαδή, στηριζόμαστε σε αυτά που υπάρχουν σήμερα, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και τις πιθανές εξέλιξεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι ήταν υπέρ των δεών επικοδομητική συζήτηση και πολύ ενθαρρυντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. <clears throat> να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κάλλας για να ολοκληρώσει τη συζήτηση και μετά θα δούμε τις προθεσμίες και νομίζω πως θα τελειώσουμε και λίγο νωρίτερα και να πιούμε και ένα καφεδάκι. Παρακαλώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας. για την παρακολούθηση του Wi-Fi, το Wi-Fi tracking. Ε, επιλογή. Όταν κάποιο βλέπει ότι παρακολουθείτε το Wi-Fi και υπάρχει ένα σήμα που το λέει, τι επιλογή έχει. Δεν μπορεί να πει δεν το δέχομαι, opt-out. Άρα ίσω έχει το αντίθετο αποτέλεσμα αν υπάρχουν αυτά τα σήματα, εφόσον δεν του δίνει καμία επιλογή. Γι' αυτό δεν το περιέλαβα. Τώρα για το πότε θα γίνουν όλα αυτά. Άκουσα τι είπατε. Και άκουσα τι είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά υπάρχει και η αντίστροφη όψη. Επειδή λοιπόν ε, θα είναι συντροματικό του GDPR οι εταιρείε, θα έπρεπε να έχουν και τα δύο, ε, γιατί πρέπει να συμμορφωθούν και τα δύο. Καλύτερα λοιπόν να τα έχουν και τα δύο την ίδια στιγμή. Όμως από την άλλη πλευρά, ότι αν είναι πολύ σύντομη η περίοδος εφαρμογής, τότε πρέπει να βιαστούν οι εταιρείε. Οπότε στη διάθεσή σας για να δούμε τι είναι καλύτερο για την ελεύθερη ροή δεδομένων βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν είμαι βέβαιη πως συνδυάζεται με το τμήμα της ε, προστασία της ιδιωτική σφαίρας για την ε, ουδετερότητα τη τεχνολογίας. Συμφωνώ ότι τα άρθρα είναι βεβαίως ε, τεχνολογικά ουδέτερα, αλλά και οι ιδεολογικές σκέψεις ε, παίζουν ρόλο, συμφωνώ. Θα πρέπει και αυτές να είναι όσο πιο ουδέτερες γίνεται. Να μην ξεχάσουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους και βεβαίως θα τα πούμε και περαιτέρω και θα συνεργαστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Ιουνίου και γνωρίζετε όλοι πως το σύστημα έχει ήδη ξεκινήσει από τις 29 ε, Ιουνίου για να έχουμε περισσότερο χρόνο προετοιμασία. αν ε, μιλάμε για το σύστημα IT4AM που μας επιτρέπει περισσότερο χρόνο για να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Ε, πάντως εδώ εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τις κελίες με το ε, χρονοδιάγραμμα των άλλων επιτροπών. Έχουμε νομίζω ένα τεταρτάκι μέχρι να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε κάπου καθυστέρησα, αλλά ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Ας αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ας κάνουμε μία ψηφοφορία για να ελέγξουμε τη λειτουργία του σύστημα. Άρχεται. I close the vote. Πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εντάξει, λειτουργεί το σύστημα. No, no, another one. Who has got you? Relax. Presidente. Sorry, sorry, small break. Two without the Ωραία, μπορούμε να αρχίσουμε. Τελικός κατάλληλος οφοριών. Διαδικαστικό. Μου φέρνουν τώρα την ε, ηλεκτρονική μου κάρτα. Ε, αλλά εάν υπάρχει κάποια αμφίροπη ψηφοφορία θα ψηφίσω όπως και η ομάδα μου. Ευχαριστώ πολύ. πρώτη έκθεση Ζωρίνιο πρόταση κανονισμού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τροπολογεί τους κανονισμούς ε, που αφορούν την προώθηση της εσωτερικής, της ε, επιγραμμικής συνδεσιμότητας ε, στις τοπικές κοινωνίες. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται και συγχαίρουμε τον εισηγητή Κρέλ στρατηγική διαστήματος για την Ευρώπη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά έλεγχος πέρας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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 18α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 και ε, μεταφορών 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Την 156. Πέρας. Αγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και την 157. 157. Πέρας. Απορρίπτω. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 162. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 Α, έχει αποσυρθεί από τους συντάκτες. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή τραν 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή ίνκο 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή πες α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πες β υπέρ κατά αποχές δεκτή πες σ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο α υπέρ κατά. Άσα ελέγξουμε. Ήμκο α. Ήμκο Α ε. Α. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά Ασέλεξουμε την 6 Ελέγχουμε την τροπολογία 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με πολύ ευρία πλειοψηφία και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Περνάμε στην επόμενη έκθεση της Αγγέλικα Μλίνερ για την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων. Τροπολογία 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2α υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 2α. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από κοινού τρεις τροπολογίες 108, 109 και 110 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 3. Και παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Δεν μπορώ να καταλάβω το αποτέλεσμα αλλιώς. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138 υπέρ 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 140, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 145 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 146 και 147 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 151. Τροπολογία 151. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 151 και επαναλαμβάνω να σηκώνετε τα χέρια σας. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 για το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον. Ας το ελέγξουμε όμως καλύτερα, γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Σας παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. 18 τμήμα 2 και πάλι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 28 πάμε στην συμβαστική 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 και 48 μαζί υπέρ. Κατά. Άποχες Απορρίπτονται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 και 73 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 74 και 75 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 74 και 75 μαζί είπα. Α, όχι, εγκρίνονται. Ε, ναι, εγκρίνονται, εγκρίνονται. Συμβιβαστική τροπολογία 13. Ήθελα να σας τσεκάρω. Τροπολογία 13, συμβαστική. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συνολική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διαδικαστικό από την κυρία Μλίναρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε παρά τη διάσταση απόψεων μεταξύ μας. Και η τελική έκβαση, το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται ούτε στην προσωπική μου ομάδα, ούτε στην ε, θέση της ομάδας μου. Ε, θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από τον τίτλο της γνωμοδότησης λόγω διάσταση από τις απόψεις μου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα αφαιρέσουμε το όνομά σας. Οπότε θα υποβληθεί ως γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας Ήτρε και όχι ως γνωμοδότηση Μλίναρ. Και θα υποβληθεί στην καθήλη αρμόδια επιτροπή ως γνωμοδότηση επαναλαμβάνω της Επιτροπής Ήτρε χωρίς να αναφέρεται το όνομα της ε, γνωμο... συντάκτηρης γνωμοδότησης. Κρίμα, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τελευταία ψηφοφορία της γνωμοδότησης του κυρίου Βέρνερ Λάγκεν. Ε, σύστημα εμπορίας εκπομπών για την αεροπορία. Τρεις τροπολογίες 40, 43, 30 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 35 άρχεται η ψηφοφορία 35, τροπολογία 35, τέλος ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 36, ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος και για αυτήν. 36, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, αυτή εγκρίνεται. 44. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 46. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες μαζί. 50, 53, 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τέλεια, μπράβο. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50... 5, συγγνώμη. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 55. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται η τροπολογία 7. 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος και πάλι. Συγγνώμη. Άρχιτη ψηφοφορία για την 3. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 12. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 15 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 17 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 18. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 ή μάλλον 21. 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 28, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Μα δεν ψηφίζεται. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα δεν βλέπω τίποτα. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 33. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 34. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Υπέρ της 4 παρακαλώ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται. Άρα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία. Άρα απορρίπτεται. 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. να την ελέγξουμε και αυτήν. 37 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Και πάλι ελέγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 ε, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική κλίση, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Και τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 51 ψήφους υπέρ και 5 κατά. Συγχαρητήρια στον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Λάγκεν. Και τώρα περνάμε στην τελευταία μας γνωμοδότηση. Συμβολή της Επιτροπής Ήτρες στο ψήφισμα της Επιτροπής ΕΜΒΗ για την COP23. Λοιπόν, θέλει κάτι να πει η Γκουέ? Όχι. Γκουέ, έχω μία υπογραφή ότι η Γκουέ συμφωνεί με τη συμβιβαστική. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Στηρίζει τη συμβαστική μας. Αν την υπερψηφίσουμε βεβαίως. Μία μόνο ψήφος είναι, ψηφοφορία, ηλεκτρονική, ε, άρχεται. Γνωμοδότηση κόπου 23. Πέρασε. Ωραία. 52 υπέρ, 4 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν όλοι εδώ. Ευχαριστώ και για τα γυαλιά. Ε, με σώσατε. Σον, εσύ κατάλαβες, είδες τίποτα ή τίποτα απολύτως. can I keep it? Μου τα χαρίζεις, να τα κρατήσω. Α, όχι, όχι για πάντα. Για σήμερα. Αγαπητοί φίλοι, τελειώσαμε νωρίτερα, 15 λεπτά. Έχουμε 15 λεπτά διάλειμμα. Γιατί στις 11 θα ξεκινήσουμε την κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Σε 17 λεπτά. Ήμασταν φοβερά γρήγοροι και αποτελεσματικοί.